herr präsident! λοιπόν άρχεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χτεσινής συνεδρίασης ε, είναι στη διάθεσή σας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που έχει αντίρρηση. Από ό,τι βλέπω όχι, ως εκ τούτου εγκρίνονται τα πρακτικά. Πάμε τώρα